Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρίσω την επανάληψη της περίοδου της Συνόδου που διεκόπη στις 29 Μαρτίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ διότι σήμερα μπορούμε να καλωσορίσουμε για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 12 Κροάτες παρατηρητές.